των νέων διορισμών θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά και εφόσον δεν εκφραστούν αντιρρήσει στους διορισμούς αυτούς θα θεωρηθούν οι διορισμοί αυτοί ότι επικαιρώνονται.